Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ε, παραλαμβάνεται λοιπόν η συνεδρίαση. Θα ξεκινήσουμε μια ανακοίνωση. Η ψηφοφορία αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου χωριστεί σε διάφορες ε, περιόδους όπως έχουμε ήδη πει δεδομένου το αριθμού των τροπολογιών και δεδομένου του αριθμού χωριστών ψηφοφοριών αυτά ε, όσον αφορά τις ε, ψηφοφορίες πληροφορίες αυτές υπάρχουν ούτως ή άλλως στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο κομμάτι το οποίο ε, λέει πληροφορίε πληροφορίες ε, και αν ε, δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση εγκρίνονται αυτές οι αλλαγές οπότε αύριο θα γίνουν τρεις γύροι ψηφοφορίας και περνάμε τώρα στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Τραπεζική Ένωση. Παράγραφος 3 εγκρίνεται. Παραγραφός 4 μέρος 1 εγκρίνεται. Παραγραφός 4 μέρος 2 εγκρίνεται. Παραγραφός 5 μέρος 1 εγκρίνεται. Παράγραφος 5 μέρος 2 εγκρίνεται. Παράγραφος 5 μέρος τρίτο εγκρίνεται μετά τροπολογία 10 στην παραγραφό 7 εγκρίνεται τροπολογία 11 εγκρίνεται που αφορά το κείμενο μετά το άρθρο 9 Παράγραφος 10 μέρος πρώτο εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο εγκρίνεται. Παραγραφός 10 μέρος τρίτο εγκρίνεται. Παραγραφός 11 μέρος πρώτο εγκρίνεται. Παράγραφος 11 μέρος δεύτερο εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Τροπολογία 5.1 εγκρίνεται. Τροπολογία 5 μέρος δεύτερο απορρίπτεται. Τροπολογία 2 απορρίπτεται. Άγραφος 14 μέρος πρώτο εγκρίνεται. Παραγραφός 14 μέρος δεύτερο εγκρίνεται. Παραγραφός 15 μέρος πρώτο εγκρίνεται. Παραγραφός 5 μέρος δεύτερο εγκρίνεται. Παραγραφός 18 μέρος πρώτο Εγκρίνεται. Παράγραφος 18 μέρος δεύτερο. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18 μέρος τρίτο. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18 μέρος τέταρτο. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 στην παράγραφο 21 απορρίπτεται. Τροπολογία 30 απορρίπτεται. Παράγραφος 31 μέρος πρώτο δεκτή. Παράγραφος 31 μέρος δεύτερο δεκτή. Τροπολογία 3 στην παράγραφο 33 απορρίπτεται. Τροπολογία 7 στην παράγραφο 36 Επίσης απορρίπτεται. Τροπολογία 12 στην παράγραφο 41 δεκτή. Μετά η 41 μέρος πρώτο καταπίπτει. όπως και το μέρος δεύτερο της παραγράφου 41 παραγραφός 44 δεκτή τροπολογία 8 για την παράγραφο 41 απορρίπτεται παραγραφός 50 απορρίπτεται παραγραφός 51 μέρος πρώτο εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο επίσης εγκρίνεται. Μέρος τρίτο της 51 εγκρίνεται. Παράγραφος 52 εγκρίνεται. Και παράγραφος 53 εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Μετά την παραγωγή 56 το Τροπολογία 9. Στο εκτιμώντας C εγκρίνεται. Και τροπολογία 1. Μετά το εκτιμώντας H Απορρίπτεται. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση περνάμε τώρα στα αποτελέσματα που σχετίζονται με τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για τον προεπιλογισμό του 2021. Τα βλέπετε ήδη στην οθόνη τα αποτελέσματα. Θα τα πούμε και λεπτομερώς. Παρουσιάζουμε μόνο τα τελικά αποτελέσματα. Τροπολογία 24. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 μέρος πρώτο. Απορρίπτεται. 8 μέρος δεύτερο. Α, απορρίπτεται. τοπολογία 9. Απορρίπτεται. 10. Απορρίπτεται. 11. Απορρίπτεται. 12. Απορρίπτεται. 13. Απορρίπτεται. 15. Απορρίπτεται. 7. Δεν κρίνεται. Τροπολογία 16. Απορρίπτεται. Μέρος πρώτο της παραγραφού 8. Εγκρίνεται. όπως και το δεύτερο μέρος της ε, παραγράφου 8 επίσης εγκρίνεται παράγραφος 9 μέρος πρώτο εγκρίνεται μέρος δεύτερο εγκρίνεται παράγραφος 11 μέρος πρώτο εγκρίνεται μέρος δεύτερο εγκρίνεται Τροπολογία 17. Το άρθρο 13. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Στο άρθρο 13. Απορρίπτεται. Άρθρο 13. Αρχικό κείμενο. Μέρος πρώτο εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο. Εγκρίνεται. Μετά. Τροπολογία 1. Στην στο άρθρο 17 εγκρίνεται τροπολογία 14 μετά το άρθρο 20 απορρίπτεται η 23 εγκρίνεται άρθρο 23 εγκρίνεται τροπολογία 25 απορρίπτεται. Παράγραφος, ε, άρθρο 26 μέρος πρώτο εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο και αυτό εγκρίνεται. Τροπολογία 18 στο άρθρο 27 εγκρίνεται. Άρθρο 30, μέρος πρώτο, εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο άρθρο 31. Τροπολογία 2. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Μετά τη 33. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Στην παράγραφο 38. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Απορρίπτεται. Παραγραφός 41 μέρος πρώτο. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο. Εγκρίνεται. Μετά έχουμε την τροπολογία 3 στο άρθρο 45. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 στο άρθρο 49. Απορρίπτεται. άρθρο 49 αρχικό κείμενο εγκρίνεται. Τροπολογία. 21 στο άρθρο 51 απορρίπτεται. Τροπολογία 4 στην παράγραφο 57 εγκρίνεται. Τροπολογία 5 μετά το εκτιμώντας α απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 6 μετά το εκτιμώντας β απορρίπτεται. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. όσον αφορά τις κατευθύνσεις ε, της Τραπεζικής Ένωσης. Περνάμε στην τρίτη ψηφοφορία. Πρώτα όμως θα δώσω τον λόγο στην κυρία Χολμάιερ. Παρακαλώ, λοιπόν, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. θα ψηφίσουμε για την επανάληψη των έρευνων κατά του Πρωθυπουργού της Τσεχίας για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είναι ένα ψήφισμα όλων των πολιτικών ομάδων μετά από το αποτέλεσμα του ταξιδιού της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Τσεχία ε, όπου είχαμε ως ευρήματα συστημική αδιαφάνεια δεν υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος και δεν αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Επίσης, η ελευθερία των μνημεία γίνεται όλο και πιο προβληματική και ασκείται πίεση στους υπαλλήλους. Το βασικό μήνυμα είναι ότι εάν επιβεβαιωθεί ε, σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να επιληθεί. Οι πιθανότητε είναι τρει. Να μην υπάρχουν πλέον αυτά τα συμφέροντα, να σταματήσουν οι επιδοτήσει ή αποχή από αποφάσεις που αφορούν αυτά τα συγκρόμενα συμφέροντα. Αν δεν είναι αυτό δυνατόν, ε, μπορεί να υπάρξει παρέτηση από το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε υπέρ καθώς οι επιδετήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ωφελούν όλο τον λαό και όχι κάποιους μεμονωμένους ολιγάρχες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε την τρίτη περίοδο ψηφοφορίας τώρα. η οποία ξεκινάει και πηγαίνει μέχρι τις 19 και 45. 8 παρατέταρτο. Οπότε, όπως ξέρετε, θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα ψηφοφορίας που έχουμε εξ αποστάσεως. Μπορείτε λοιπόν από τώρα, όπως είπαμε, μέχρι τις 19.45 μπορείτε να ψηφίσετε ώρα Βρυξελών βέβαια. Και στις 10 και 4 θα επανέλθουμε για τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Λίγη συνεδρίαση.